prepared for very, very uninteresting. Okay, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω. Καλημέρα σας. Ξεκινάμε για το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Έλεγχος εφαρμοστικών μέτρων και εξουσιοδότηση πράξεων είναι ένα τμήμα των αρμοδιοτήτων των ελεγκτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν θέματα λοιπόν. Να καλωσορίσω τον κύριο Μπερναρντίνο, τον νέο πρόεδρο ε, της ΕΙΟΠΑ και τον Σβεν Γκέτνερ της Αρμόδιας Επιτροπής. Θα συζητήσουμε για τα κρύψη και ιδιαίτερα τα νέα τεχνικά standards, διακανονιστικά νέα τεχνικά standards, μετά από τη δημόσια διαβούλευση θα υποβληθούν μέχρι το τέλος του μήνα ή μάλλον μέχρι το τέλος του Μαρτίου αν καταλαβαίνω καλά. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ότι και εδώ έχουμε κάτι το οποίο θα βοηθήσει πολύ την προστασία των επενδυτών στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των χρηματαγορών και θα επηρεάσει το διακανονιστικό τους πλαίσιο. Σημαντικό κομμάτι λοιπόν και αυτό της δραστηριότητάς μας. Θα τα συζητήσουμε αργότερα αυτά μετά από τις παρουσιάσεις Μπερναρντίνο και Γκέρτνερ. Η κυρία Μπερές δεν είναι παρούσα σήμερα, η Ελίσα Φερέιρα θα μιλήσει εξ ονόματός της. Θα ήθελα όμως να δώσω αμέσως το λόγο στους κυρίους κυρίους Μπερναρντίνο και Γκέτνερ για να κάνουν μια εισαγωγή όχι πάνω από 10 λεπτά και οι δύο μαζί. Γκάμπριελ Μπερναρντίνο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε όλους. Έχει μεγάλη σημασία για μας που βρισκόμαστε σήμερα εδώ για το θέμα των PRIPS. Ξέρετε ότι η προσπάθεια για το ενημερωτικό έγγραφο είναι σημαντικό για την Επιτροπή μας στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό από το 2012, είμαστε σε επαφή με πανεπιστημιακούς ερευνητές και εκπροσώπους της βιομηχανίας. Έχουμε κάνει και μία μελέτη έρευνα μάλλον σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Συμβουλευτική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων. Έχουμε φτάσει στο, στην τελική φάση μετά από το κλείσιμο της επεξεργασίας στο τέλος Ιανουαρίου. Πήραμε πάνω από 100 εκτεταμένες απαντήσεις, πολλοί εμπλεκόμενοι έχουν ζητήσει να υπάρξουν βελτιώσεις του RPS και να υπάρξει το λεγόμενο fine tuning. Το θέμα είναι πως το RTS αυτό θα περιλαμβάνει τις πολλές και διαφορετικές μορφές των PRIPS. Οι επιλογές τις οποίες έχουμε είναι μια προσπάθεια εξισορρόπησης και στάθμισης Υπάρχουν κάποια επιπλέον στοιχεία στα οποία οι απαντήσεις δεν δέχονται τις προτινόμενες από πλευράς μας ισορροπίες, αλλά είναι σαφές ότι οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες. Έχουμε περάσει πλέον στους χρονισμούς και τις ε, ρυθμίσεις για την εφαρμογή. Έχουν εκφραστεί ανησυχίες τα τελευταία χρόνια για την τελική μορφή του δεσμευτικού κειμένου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου όταν θα υπάρξει συνάντηση εκπροσώπων όλων των προϊόντων. Οι περισσότερες ε, αντιπροσωπείες ζητούν να υπάρξει μια περαιτέρω ε, θα έλεγα παράταση της περίοδου επεξεργασίας και δεχθήκαμε τους εννέα μήνες ως προς αυτό. Εμείς πάντως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη συμφωνημένη πρόταση RTS στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 31 Μαρτίου όπως είπε ο Πρόεδρος και αυτό είναι κάτι στο οποίο εμένουμε. Αλλά κατά τη διάρκεια αυτής της διαβούλευσης και ακούγοντας τα επιχειρήματα της βιομηχανικής, της, της, της επιχειρηματικής πλευράς, προφανώς κατανοούμε τις ανησυχίες και θα πρέπει να αφήσουμε χρόνο και στους Ευρωπαίους νομοθέτες. Τώρα να δούμε πού είναι τα προβλήματα τα οποία συναντήσαμε στο παρελθόν. Καταρχάς για τον κίνδυνο. Ο δείκτης για τον κίνδυνο θα είναι από τα βασικά του kit που θα προτείνουμε. Εμείς καθοδηγούμεθα από την τροφοδοσία η οποία προήλθε από το τεστ που έγιναν στους καταναλωτές. Ε, υπήρξαν ε, βαθμολογήσεις, ε, ε, υπάρχει βέβαια μια πιο περίπλοκη μεθοδολογία για την χρήση συγκεκριμένων PRIPS. Εμείς χρησιμοποιήσαμε επίσης δεδομένα ποσοτικού τύπου αλλά με ορισμένα ποιοτικά στοιχεία. Λάβαμε υπόψη μας τα διαφορετικού τύπου κρύψη τα οποία πρέπει να καλυφθούν συνολικά. Αναπτύξαμε εμείς μια μεθοδολογία υπολογισμού κινδύνου που λαμβάνει υπόψη και τις ανάγκες των περίπλοκων προγραμμάτων και εμείς περιμένουμε τις τελικές απαντήσεις στο έγγραφο διαβούλευσης. Υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με τη στάθμιση που πρέπει να προηγηθεί τη διάκριση των διαφορετικών προϊόντων. Υπάρχουν επίσης και προκλήσεις σε σχέση με την αξιολόγηση των κινδύνων των πρίξ που είναι κατασκευασμένα με σωστό τρόπο. Ελπίζουμε ότι θα δώσουμε τις απαντήσεις ε, τους επόμενους, τις επόμενες μέρες. Τώρα η απόδοση ε, είναι βασικό. Έχουμε αναπτύξει μέτρα έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε προοπτικές μορφές ενημέρωσης και πληροφόρησης για τις επιδόσεις των προϊόντων αυτών. Έχουμε εξετάσει πάρα πολλές δυνατότητες. Τα τεστ των καταναλωτών δείχνουν ότι οι καταναλωτές δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν πάντα τις προβλεπτικές αν θέλετε ε, παρουσιάσεις για τις αποδόσεις ε, των συγκεκριμένων προϊόντων. Και έτσι θα πρέπει να, να υποχρεώσουμε αυτούς που παρασκευάζουν τα συγκεκριμένα προγράμματα να ενημερώνουν με πιο απλό τρόπο. Ε, έχουμε λοιπόν προσπαθήσει να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας συνδέοντας σαν παράδειγμα τις αναμενόμενες αποδόσεις με τα επίπεδα κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα ΠΡΙΠ έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές δυνατότητες εξέλιξης. Εξετάζουμε επίσης ε, και ε, τις αποδόσεις στο παρελθόν των αντίστοιχων προϊόντων. Κάποιοι εμπλεκόμενοι μας ζήτησαν να συμμεριλάβουμε επίσης και τις καλύτερες επιδόσεις σαν χρήσιμα σενάρια. Βλέπουμε ότι τέτοιες πληροφορίες θα ήταν χρήσιμες προσθήκες εφόσον βέβαια δείχνουν τις ε, πραγματικές αποδόσεις μετά από την αφαίρεση του κόστους. Καθαρές αποδόσεις. Τώρα για τα κόστη. Γνωρίζουμε ότι πολλοί καταναλωτές δεν προσέχουν το κόστος των προϊόντων αυτών όταν αποφασίζουν να κάνουν επενδύσεις. Οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα όταν συγκρίνουν προϊόντα με διαφορετική δομή κόστους. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε λοιπόν μια μέθοδο η οποία θα επιτρέψει τη σύγκριση ανάμεσα σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα. Έχουμε κάποιους δείκτες για το άμεσο και το έμεσο κόστος ε, έτσι ώστε να δούμε ποια είναι τα μεμονωμένα κόστη ε, τα one-off όπως λέγεται τα άπαξ κόστη ή και τα κόστη τα οποία επαναλαμβάνονται μέσα σε μια χρονική προθεσμία. Έχουμε προτείνει επίσης ε, και την μέθοδο της μείωσης της απόδοσης για να διασφαλίσουμε την βέλτιστη δυνατή συγκρισιμότητα ανάμεσα σε δομές διαφορετικά για το κόστος. Έτσι θα βελτιώσουμε τη διαφάνεια και την ισοτιμία ανάμεσα στα διάφορα προϊόντα. Η ανάλυση που κάναμε εμείς τις απαντήσεις του εγγράφου ε, διαβούλευσης μας επιτρέπουν να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις αλλά όχι μείζονες αλλαγές. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε καλύτερα και την μεθοδολογία σε σχέση με τα κόστη συναλλαγής για να είναι πιο εφαρμόσιμα. Όπως επίσης ε, η παρουσίαση του κόστους στο kit πρέπει να είναι απολύτως κατανοητή. Και αυτό το είδαμε και από τις απαντήσεις και από τα τεστ που κάναμε. Ε, πρέπει να υπάρξει μια νέα μορφή εναρμόνισης ε, των μεθόδων υπολογισμού του κόστους των προϊόντων. Ε, αυτό είναι τα σωστά θεμέλια θα έλεγα για τα προϊόντα αυτά στο μέλλον. Ελπίζω να σας βοήθησα με αυτά που σας είπα και θα ακούσω και τις δικές σας απόψεις για την τελική πρότασή μας για τα RTS και τα πρίψη στο μέλλον. Ευχαριστώ αγαπητέ Μπερναρντίνο και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκάρτνερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε σήμερα εδώ. Καλωσορίζουμε την ε, πρώιμη εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την υπόθεση και την ευκαιρία που μας παρέχεται μέσω αυτής της ακρόσης να συζητήσουμε την πρόοδο και τα τελευταία βήματα που μας περιμένουν στο επίπεδο 2 του κανονισμού ΠΡΥΠΣ. Ε, έχουμε ε, να εστιάσουμε στο χρονοδιάγραμμα και την έγκριση και φυσικά με χαρά θα απαντήσω σε άλλες ερωτήσεις αν έχετε. Το πακέτο PRIPS αποτελεί ένα πραγματικά μεγάλο βήμα μπροστά στην βελτίωση της διαφάνειας των επενδυτικών προϊόντων στους διάφορους τομείς. Θα χρησιμοποιηθεί από τους καταναλωτές σε καθημερινή βάση, ώστε να προβαίνουν σε ενημερωμένες αποφάσεις περί επενδύσεων. Είναι επίσης μια πρωτοβουλία που θα είναι άμεσα ορατή στους πολίτες της Ένωσης. Πραγματικά λοιπόν εδώ πρέπει να τα καταφέρουμε. Ε, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι δεσμευμένα να ανταποκριθούν στην, ε, χρονο, ε, προθεσμία για την εφαρμογή του ΠΡΙΠΣ και η Κομισιόν συνεργάζεται πλήρως με τις τρεις ΕΖΑ εποπτικές αρχές και έχει ζητήσει και νομικές συμβουλές σε σχέση με την ερμηνεία του κανονισμού κάθε του μορφή. Ε, επίσης, για να είναι πλήρως ε, κατανοητό και πραγματικά χρήσιμο για τους επενδυτές, η Κομισιόν έχει προβεί σε έλεγχο των, μια δοκιμή μάλλον με τους καταναλωτές, που θα καταλήξει στην τροφοδότηση με πληροφορίες του ίδιου του πακέτου. Αυτή τη στιγμή που θα έχουμε τη γνωμοδοτήση των εποπτικών αρχών, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε στο RTS πριν το καλοκαίρι, ώστε να έχουν οι νομοθέτες το χρόνο να ασκήσουν το δικαίωμα ελέγχου τους. Ξέρουμε ότι κάποιες δοκιμές μπορεί να καθυστερήσουν την νομοθεσία, ε, την εφαρμογή μάλλον της νομοθεσίας πρίψης, λόγω του ότι θα ισχυριστούν ότι δεν έχουν το χρόνο να προσαρμόσουν τα συστήματά τους. Είναι φιλόδοξο το σχέδιο, όμως από τη στιγμή που θα υποβληθεί το RTS στα τέλη του Μαρτίου στην Κομισιόν μέχρι την εφαρμογή του στις 31 Δεκεμβρίου ε, θα είναι δύσκολο αλλά θα είναι δυνατόν ο κλάδος να προετοιμαστεί. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στις συμπεφωνημένες ημερομηνίες γιατί είναι εφικτό και είναι σημαντικό το πακέτο αυτό να είναι διαθέσιμο και άρα οι καταναλωτέ να έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε να προβούν στις επενδυτικές τους αποφάσεις να μιλήσω για δύο συγκεκριμένα θέματα. Όσον αφορά την ε, ανάθεση στην Κομισιόν για να μπορέσει το πρίψη να στοχεύσει συγκεκριμένους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς ε, στόχους. Ο Επίτροπος Χίλε μας ανέθεσε να προετοιμάσουμε μια συμβουλή για τις υποπτικές αρχές που θα εστιάζει στις συγκεκριμένες διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι κατασκευαστές των πρίψ στοχεύοντας σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους. Όμως για να μην ε, ε, αποτραπούν οι στόχοι περιορισμένοι των ΕΖΑ, οι πόροι περιορισμένοι των ΕΖΑ, ε, θα πρέπει αυτό να γίνει από τη στιγμή που το πακέτο θα έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, οι αρμοδιότητες πρόληψης υπό την ε, ΜΥΦΙΡ, από τις Εθνικές Αρχές, έχουν αποδεσμευθεί οι διάφορες αρχές και αυτό σύμφωνα με την νέα διοργανική συμφωνία που δεν επιτρέπει την τραπεζική διαδικασία και τις αποφάσεις ε, να λαμβάνονται από δύο διαφορετικές αρχές. Άρα λοιπόν το ΠΡΙΠΣ θα είναι πλήρως εναρμονισμένη από την 1η Δεκεμβρίου 2016. Η υιοθέτηση και εφαρμογή ε, των παρομοίων αρμοδιοτήτων υπό την ΜΥΦΙΡ θα υιοθετηθούν στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο της Μηφύρα. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Και τώρα λοιπόν να ακούσουμε και τις παρεμβάσεις των μελών. Εξ ονόματος ε, του εισηγητή η Ελίζα Φεραίρα. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Βερέση, η εισηγήτρια ζητά συγγνώμη, αλλά δυστυχώ δεν μπορέσει να παραπληθεί εδώ σήμερα. Άρα θα μιλήσω εγώ για αυτήν. Να ευχαριστήσω και τους δύο προηγούμενους ομιλητές για τις πληροφορίες που μας έδωσαν. Κάποιες εξ αυτών καλύπτουν κάποιες από τις ερωτήσεις που θέλαμε και εμείς να υποβάλουμε. Θα θέλαμε ωστόσο να έχουμε και πιο πολλές πληροφορίες για τις επόμενες ερωτήσεις. Πρώτο σχόλιο. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Επειδή ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση από τις υποπτικές αρχές, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα το προβλεπόμενο. Καλώς ορίζουμε το γεγονός ότι και οι δύο προλαλήσαντες μίλησαν για το χρονοδιάγραμμα. Και επιτέρως ε, η ημερομηνία της 31 η Μαρτίου που ανέφερε η ΙΟΠΑ. Συνάδει αυτό με την προθεσμία τέλη Ιουνίου που είχαμε κατά νου. Προκειμένου λοιπόν να έχει επαρκή χρόνο και το Κοινοβούλιο και, η... ο οικονομικός κλάδος. Τώρα, για κάποια συγκεκριμένα θέματα, αυτό που έθεσε και ο κύριος Μπερναντίνο, αλλά μας ε, απασχολεί το θέμα του πώς οι υποπτικές αρχές και ιδιαίτερα ο ΑΕΟΠΑ προτίθενται να αντιμετωπίσουν τη διατύπωση στο επίπεδο 1 για τα κατάλληλα σενάρια. Κοιτώντας τι έχει γίνει στο παρελθόν, μπορεί απλά να παραταθούν κάποιες τάσεις. σε ό,τι αφορά τα αισιόδοξα σενάρια, πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο θα συνεχιστούν οι τάσεις αυτές ο κ. Μπερναντίνο είπε ότι θα γίνει αν ε, ισχύσει αυτό. Αλλά μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτές τις προβλέψεις. Είναι ένα σημείο κριτική στην ανάλυση και στην αξιολόγηση κινδύνου. Θα θέλαμε λοιπόν να μάθουμε πιο πολλά στοιχεία γι' αυτό. Καλωσορίζουμε επίσης την πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής να να το μύθι και το Όχι μόνο στην ΑΙΟΠΑ, αλλά και στις εποπτικές αρχές, για να τις ενισχύσει. Και οι εξουσίες ε, επέμβασης των υποπτικών αρχών θα πρέπει να περιγράφονται με σαφέστατο τρόπο. Ένα τρίτο στοιχείο. Ε, δουλεύουμε με συγκεκριμένους ε, δείκτες και το πόσο ερμηνεύουμε τους δείκτες αυτό αποτελεί ένα αυθαίρετο στοιχείο από μόνο του. Ωστόσο, ο τρόπος ε, καθορισμού των δικτών καλωσορίζει, ε, μάλλον καθορίζει και την αντίληψη του ρίσκου, του κινδύνου. Εξηγήστε μας λοιπόν αυτό το τεχνικό έργο που κάνετε για να συνοψίσετε τους δείκτες χωρίς να χάσετε σημαντικές πληροφορίες. Επίσης θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει στις εποπτικές αρχές δυνατότητες αξιολόγηση όλων των χρηματοδοτικών μέσων σε ό,τι αφορά και τα τρίπ, σε ό,τι αφορά τα δεδομένα τα οποία θα πρέπει να δίδονται σε περίπτωση πολλαπλών δυνατοτήτων επενδύσεων. Πέμπτη ανησυχία για τα παραγωγά. Τα λόμπι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα εξαιρεθούν από το πέντε εφαρμογή. Αυτό το καταπολέμησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερο συγχαίρη ήταν και η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Τελευταίο σημείο για την φορολογία. Δεν συμπεριληφθήκε το το 1 το πρίψ. η φορολογία. Είναι επίση σημαντικό σε ό,τι αφορά την απόφαση ε, επενδύσεων. Να δούμε πώς θα το χωρέσουμε, πώς θα μπει στην αξιολόγηση. Αυτά επί του παρόντος. Και φυσικά θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερες προσθέτε πληροφορίες από την ΕΟΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την προσέγγιση και τον διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. τι κάνουν από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους δύο ομιλητές για τις ε, πολύ ακριβές πληροφορίες που μας έδωσαν, πολύ χρήσιμες από την ε, συζήτησή μας. Και όντως απάντησαν ήδη κάποιες ερωτήσεις που έχουμε. Ένα κρίσιμο στοιχείο για το Κοινοβούλιο, για όλο το Κοινοβούλιο μάλιστα, όταν συζητήθηκε, είναι το να μην υπάρξει καθυστήρηση να μην υπάρχει καθυστέρηση ό,τι αφορά τι πραγματικέ ε, αρμοδιότητε, ε, ακόμα και αν καθυστερήσει το MIFID, και να υπάρχουν ε, σωστέ και κατάλληλε δυνατότητε παρέμβαση να προβλεφθούν. Έχουμε πληροφορίε ότι δεν θα ισχύσει όμω κάτι τέτοιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά δηλαδή την έγκυρη εφαρμογή. Ένα δεύτερο στοιχείο. Σε ό,τι αφορά τον ε, δείκτη κινδύνου. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτόν τον δείκτη, Πρέπει να σας πούμε ότι διαφέρουν τα επίπεδα σε ό,τι αφορά τους επενδυτές. Και έτσι λοιπόν ε, ε, τα διαφορετικά επίπεδα ανάλογα και με το επίπεδο εκπαίδευσης του καθενός. Αλλά ε, για αυτούς που έχουν διαφορετικό επίπεδο θα είναι δύσκολο να υπάρξει και σύγκριση των παραγόντων κινδύνου και θα πρέπει να ξανακοιτάξουμε την μεθοδολογία τι μέθοδο που θα εφαρμόζονται. Καταρχά. Πώς οργανώνονται και μία διαδικασία αναθεώρησης, αξιολόγησης για να δούμε αν λειτουργεί σωστά. Ύστερα, με ικανοποίησαν τα σχόλια σε ό,τι αφορά το κόστος. Ήταν ε, η θετική απάντηση που δόθηκε για ότι θα υπάρξει ένα γράφημα για τους δείκτες και για τον αντίκτυπο, ε, για την απόδοση σε ό,τι αφορά το πραγματικό κόστος και τη μείωση της απόδοσης. Δεν ήταν σαφές όμως σε ό,τι αφορά το κατά πόσο θα αναφέρεται το σωρευτικό αντίκτυπο του κόστου στους δείκτες αυτούς. Αυτό θα μπορούσε να αποβεί δύσκολο, ξέρετε, για ένα τμήμα των καταναλωτών. Γιατί μπορεί να είναι και ηλικιωμένοι, για παράδειγμα, οι καταναλωτές αυτοί. Υπάρχει ένα 2% του κόστους, 8% του κόστους. Είναι δύσκολο να βρούμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος μακροπρόθεσμα, μακροπρόθεσμες επενδύσεις και προφανώς σωρευτικά μπορεί να αποτελεί αυτό ένα σημαντικό τμήμα του ίδια της απόδοσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την απόδοση κατά το παρελθόν και την παράταση των τάσεων, ήταν σαφές το κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά το σημείο αυτό, ακούσαμε πολλούς εμπειρογνώμονες του κλάδου σε ό,τι αφορά την παρελθοντική απόδοση, είτε πρόκειται για παράταση στο μέλλον, είτε όχι θα ήταν ενδιαφέρον ε, ενδεχομένω για κάποιου οικονομικού κλάδου. Δεν είμαι όμω πεπισμένη ότι είναι προ το συμφέρον των ε, καταναλωτών και επενδυτών. Γιατί όπω ξέρουμε αυτό δεν αποτελεί καμία εγγύηση για το μέλλον. Δεν υπάρχει καμία γραμμική εξέλιξη και μπορεί να είναι εξαιρετικά παραπλανητική αυτή η τάση και υπάρχουν και περιπτώσεις όπου υπάρχει ένα πακέτο το οποίο δεν τα πήγε καλά στο παρελθόν. Μπορεί να κλείσει λοιπόν ενδεχομένω ε, ο φάκελο αυτό και να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Και ω εκ τούτου λοιπόν αυτό το καινούριο στοιχείο να είναι πολύ πιο παραπλανητικό. Γιατί θα προδιαγράψει μια μελλοντική τάση θετική ενδεχομένω. Επ' αυτού λοιπόν θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας. Άλλα δύο στοιχεία. Το θέμα του πεδίου εφαρμογή. Θα ήθελα να ακούσω μια οριστική απάντηση κατά πόσο οι ανταλλαγέ και συναλλαγέ στα παράγωγα συμπεριλαμβάνονται ή όχι. Και ό,τι αφορά, τους, ό,τι δείκτες για το περιβάλλον. Πώς θα συνδεθούν με τους δείκτες ανάπτυξης που βρίσκονται υπό κατάρτιση στον ΩΣΑ και περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία για την καθολική αναφορά της Eurostat. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να είναι κοινοί αυτοί οι δείκτες κινδύνου με αυτούς άλλων κλάδων. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την πληροφορίε και πολύ λυπάμαι δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ γιατί έχω άλλε υποχρεώσει ανηλυμένε, αλλά θα φροντίσει ο βοηθό μου να σημειώσουν τι απαντήσει σα και σίγουρα θα τι λάβω υπόψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Βήμα, για το ECR. Σα ευχαριστώ όλου που θέσατε τα θέματα. Θα μιλήσω εξ ονόματος του σκιώδους εισηγητού της ομάδας μου, του Σαΐτ Καμάλ. Ε, βέβαια και εγώ έχω ασχοληθεί με το ΜΥΦΙΔ, οπότε κατανοείτε γιατί θέση. Τέσσερα θέματα θέλουμε να θέσουμε, ίσως κάποια να έχουν τεθεί από συναδέλφους. Καταρχάς, επιπτώσεις της καθυστέρησης μύφων, προηγούμενες αποδόσεις, πολλαπλές επιλογές και επίσης ε, τι ακριβώς γίνεται με τα παράγωγα. Λοιπόν, οι καθυστερήσεις ε, για το MIFID θα επηρεάσει τα PRIPS στα πλαίσια των κανόνων προστασίας των επενδυτών. Είναι αναπόφευκτη η καθυστέρηση, αλλά αυτός που φτιάχνει ένα kit στα πλαίσια του PRIPS δεν θα έχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να είναι ε, συμβατές με το MIFID 2. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε λίγο περισσότερη ε, διαφάνεια, λίγο περισσότερη ευκρίνεια, ε, πώς δηλαδή ουσιαστικά να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της καθυστέρησης. Τώρα, ε, να υπογραμμίσω το θέμα της συμπερίληψης της προηγούμενης απόδοσης ή των προηγούμενων αποδόσεων. Εδώ διαφοροποιούμεθα από άλλους συναδέλφους. Και οι δύο πλευρές βλέπω ότι θέλουν να προσθέσουν τις προηγούμενες αποδόσεις. Αυτό είχε συζητηθεί στο ε, level 1 και έχει αρχίσει να συζητάτε και στα πλαίσια του level 2. Είναι σημαντικό γιατί η απουσία των στοιχείων προηγούμενων αποδόσεων είναι ζημιογόνος. Κατανοούμε βέβαια ότι θα πρέπει να αποφασιστεί μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος και δεν μπορεί να υπάρχει λογική pick and choose και θα πρέπει επίσης να είναι συγκεκριμένη και η αναφορά σε ένα προϊόν αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε τη διαχείριση των ταμείων από τις προηγούμενες αποδόσεις τους τώρα στις πολλαπλές επιλογές επενδύσεων. Ε, ο Σαΐντ θεωρεί ότι το kit για τα πρίψ θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο αυτού του τύπου των επενδύσεων. Αλλά οι εξαιρέσεις για μέχρι το 2020 θα επιτρέψουν στους managers να καλύψουν τις συνέπειες των καθυστερήσεων. Η ομάδα μας όμως ανησυχεί για τις προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει σε σχέση με το level 2. Η ιδέα ότι μπορεί οι διαχειριστές σαν παράδειγμα να παράγουν οι ίδιοι σε εθελοντική βάση ένα kit ενημερωτικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι ε, συμβατό με την σωστή κυκλοφορία των kit ε, για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Και τέλος θέλω να υπάρξει ε, σωστή ενημέρωση σε σχέση με τα εμπορικά παράγοντα και τις ανταλλαγές των παραγόγων. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο άπτεται άμεσα των PRIPS, ε, αλλά κάποιες εμπορικές, απλές, απλά εμπορικές συναλλαγές θα πρέπει να μην θεωρούνται σαν πλήρη ε, προϊόντα και γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο. Ευχαριστώ, Κέι. Για τους φιλελεύθερους, Γιέτσκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να επαναλάβω αυτά τα οποία ακούστηκαν για τις επενδυτικές, πολλαπλές επενδυτικές δυνατότητες, επιλογές πρέπει να δοθούν καλύτερες απαντήσεις επίσης ε, γύρω από την προετοιμασία των ΚΙΤ. για τα σενάρια των προηγούμενων αποδόσεων έγιναν κάποιες συζητήσεις στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της δυνατότητας εφόσον βέβαια περιλαμβάνει ένα μείγμα πολλαπλών σεναρίων που ε, με τη σειρά τους συμπεριλαμβάνουν και τις παλαιές αποδόσεις. Thank you. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ε, για την ΚΟΕ που θα ήθελε το λόγο. Ούτε και από πλευρά των Πρασίνων δεν υπάρχει κάποιος ομιλητής. Θα ξεκινήσουμε το Catch the Eye. Ο Φέρμπερ έχει ζητήσει το λόγο. Ε. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για την ε, παρουσίαση σε ό,τι αφορά την διάμεση κατάσταση. Δεν μιλάω αγγλικά, αλλά έχουμε διαμηνία. Κοίταξα το ε, έγγραφο εργασία των τριών επιπτικών αρχών σε ό,τι αφορά το βασικό κόστο και όλα τα στοιχεία αυτά. Τα εξέτασα με προσοχή και σα απέστειλα και ε, ε, γραπτά σχόλια στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ. Πιστεύω ότι ιδιαίτερα ο κίνδυνος, ο δείκτη του κινδύνου μπορεί να αποτελέσει ένα βασικότατο στοιχείο του εγγράφου αυτό, γιατί οι πιο πολλές μελέτες υποδεικνύουν ο τελικός χρήστης και αυτός μας απασχολεί στην τελική ανάλυση δύσκολα μπορεί πραγματικά να ρυθμίσει τον κίνδυνο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και είτε υποτιμά τον κίνδυνο πριν το 2008 ή τον θεωρεί πολύ πιο μεγάλο από την πραγματικότητα σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα. Το βασικό λοιπόν είναι το πώς μπορούμε να δώσουμε στον καταναλωτή τόσο, τόσο πολλές πληροφορίες ώστε να μπορεί ενημερωμένο να λάβει μια σωστή απόφαση, να υπάρχει ένα ειδικό τέτοιο δείκτη. Αυτό ο δείκτη λοιπόν θα πρέπει να τα έξι στοιχεία. Καταρχά, τι θα πρέπει να υποδεικνύει αυτό ο δείκτη, αυτό ο θεμελιώδη δείκτη, πόσο υψηλό είναι ο κίνδυνο συνολική ζημία με ένα γράφημα. Να μπορεί να καταλάβει και ο μέσο ε, πελάτη με μία κλίμακα 0 100, όχι 1 7, τι γίνεται και θα πρέπει να μπορεί να είναι συγκρίσιμος ο δείκτης αυτός για διάφορες κατηγορίες. Να είναι ανεξάρτητος, δηλαδή να μην έχει να κάνει με τον παραγωγό ή τον έμπορο, την εμπορία του προϊόντος και θα πρέπει ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να παρακολουθεί την ε, εξέλιξη του κινδύνου του προϊόντο. γιατί ενδεχομένω κάποια άλλη στιγμή, μάλλον μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, είναι διαφορετικό ο κίνδυνο σε σχέση με δύο χρόνια μετά. Γιατί οι ειδικοί επενδυτέ είναι μακροπρόθεσμοι στι επενδύσει του. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα παρακολούθηση τη εξέλιξη του προϊόντο. Θα πρέπει λοιπόν τα κριτήρια αυτά να έχουν την προστατεύμένη αξία. Μιλήσατε λοιπόν για την εισαγωγή ε, ενός ε, παράγοντα κινδύνου της αγοράς γιατί να για τις εξελίξεις και τις ε, διακυμάνσεις στην αγορά. Δεν ξέρουμε κατά πόσον για τον ιδιωτικό επένδυτη είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο και το ίδιο ισχύει και για την ε, δίκτυα. Ε, για την ε, εκτίμηση των ε, πίστασεων. Σε ό,τι αφορά την κλίμακα 1-7, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χοντροκομμένη. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ 3 και 4 και δεν ε, υπάρχει πραγματικά εγγύηση για την ανεξαρτησία του δίκτυ. Ρωτώ λοιπόν, υπόστηρίζετε τα στοιχεία αυτά τα οποία προτείνω και πώ θα μπορούσατε να τα εντάξετε στο έγγραφο εργασία σα. Thank you. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Θέλω και όπως οι υπόλοιποι να σας ευχαριστήσω για τι εισηγήσεις. Συμφωνώ με όλου του συνάδελφου ότι πρόκειται για πολύ σημαντική νομοθεσία για την προστασία των επενδυτών. Και Θεωρώ ότι είναι κομμάτι του CMU. Θέλουμε να έχουμε περισσότερες λιανικές επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Είναι σημαντικό οι επενδυτές να εμπιστεύονται αυτά τα εν λόγω προϊόντα. Και αυτό βέβαια οδηγεί στο έλλειψη κρυφού κόστους και στη διαφάνεια στη σύσταση αυτών των επενδυτικών προϊόντων. Η νομοθεσία ε, πρώτου επίπεδου καθιστά αυτή την παρατήρηση πολύ σαφή και είναι σημαντικό να φτιάξουμε σωστά και την δεύτερο επίπεδου νομοθεσία. Και αν αυτό εφαρμοστεί σωστά από το τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι κανόνες θα είναι απόλυτα σαφείς. Εγώ έχω κάποιες ανησυχίες για σε διάφορες προσεγγίσεις ε, και τα διάφορα σενάρια απόδοσης ε, που παρουσιάζουν στους επενδυτές, δηλαδή τις, ε, τα δυνητικά τους κέρδη από αυτή την επένδυση. Εάν δώσουμε εξαιρετικά μεγάλη ευελιξία στους παραγωγούς να επιλέγουν εξαιρετικά αισιόδοξα σενάρια, Μπορεί αυτό να φανεί επικίνδυνο. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να ζητήσουμε να υπάρξει μια πολύ πιο συγκεκριμένη προσέγγιση όσον αφορά την επιλογή των σενάριων απόδοσης. Καλωσορίζω την το, απέτηση υπό το πρίψο ότι όλα τα αριθμιστικά κόστη θα πρέπει να είναι φανερά. Γιατί πολύ συχνά υπάρχουν κρυφά κόστη, όπως το κόστος συναλλαγής, που τελικά αφαιρείται από την αξία του, της επένδυσης. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι δυνατόν να γίνει η αποκάλυψη αυτή του κόστους όσο γίνεται πιο εύκολη για τους ε, καταναλωτές. Το κόστος και η μείωση της απόδοση θα πρέπει να ε, σημειώνονται με αριθμούς και όχι με ποσοστά και φυσικά ο τομέα λέει ότι ανησυχεί για το κόστος και το κόστος τη διαφάνεια, αλλά εγώ πιστεύω πω είναι εξαιρετικά σημαντικό εάν δούμε τι κάνουμε αλλού όπω α πούμε στην οδηγία ε, για, τους, για την κερδοσκοπία είναι σημαντικό να έχουμε σαφείς πληροφορίες για το κόστος χωρίς να υπάρχει υπερβολική πληροφόρηση. Πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη κατανομή του κόστους για να συμπεριληφθεί και η διαφάνεια. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει οι επενδυτές, αυτοί οι μικροί επενδυτές να μπορούν να έχουν όσο γίνεται μεγαλύτερη διαφάνεια πριν επενδύσουν. Thank σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλον. Ο Γκαμπριέλ Μπερναρδίνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας. Εκφράσατε τις ανησυχίες σας και πιστέψτε με είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποια είναι τα βασικά προβλήματα και ανησυχίες. θα προσπαθήσω να καλύψω όλα τα θέματα και να κλείσω στο τέλος. Για το χρονοδιάγραμμα και ένα δύο το αναφέρεται αυτό και όπως έχω πει και παλιότερα θέλω να με σαφής. Θα, θα επιμείνουμε σε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Αυτό είναι βέβαιο. Έχουμε ετοιμάσει τα πάντα, βεβαίως και τη δουλειά που κάνουμε στο επίπεδο της Μικτής Επιτροπής ε, και με τα τρία συμβούλια των τριών υποπτικών αρχών, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε έτοιμο στα τέλη Μαρτίου το δικό μας ε, κομμάτι. Αυτό είναι ο στόχος και σε αυτό θα επιμείνουμε. Τώρα, η την απόδοση και τα κατάλληλα σενάρια ε, απόδοσης. Εξετάζουμε αυτές τις καταστάσεις με τρία διαφορετικά σενάρια, τρει διαφορετικές υποθέσεις με διάφορες προεκβολές για το μέλλον. Φυσικά αυτό μας πήρε κάποιο χρόνο για να τα τελειοποιήσουμε. Υπήρξε ένα επιχείρημα στη διαβούλευση και αναφέρθηκε και από εσά ότι δηλαδή η υπερβολική ευελιξία που έχουμε εδώ περιλάβει μπορεί να είναι προβληματική. Αυτό το έχουμε λάβει υπόψη μετά από τη διαβούλευση και τώρα εργαζόμαστε για αυτά τα τρία διαφορετικά, τις τρεις διαφορετικές υποθέσεις έτσι ώστε να δώσουμε περισσότερα λεπτομέρειες. για το πώς αυτές οι υποθέσεις επί των οποίων βασιζόμαστε θα λειτουργήσουν. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την απόδοση. Υπάρχει και αυτό το θέμα της προηγούμενης απόδοσης. Βέβαια, η προηγούμενη απόδοση δεν είναι απαραίτητο δείκτης για το μέλλον και μπορεί να είναι και παραπλανητική και γι' αυτό θέλαμε να ακούσουμε και τις θέσεις σε αυτό. Ε, καλό θα ήταν κατά τη γνώμη μας να υπάρχει ένας συνδυασμός των ε, προβαλόμενων υποθέσεων με τις ε, προηγούμενες αποδόσεις. Γιατί θα πρέπει να είμαι ειλικρινής. Αυτό που ακούω από τους από τον τομέα είναι ότι ο κόσμος ψάχνει να βρει δείκτες για την προηγούμενη απόδοση και είτε δεν υπάρχουν, είτε εάν υπάρχουν δεν μιλάνε για την πραγματική απόδοση. Και τότε υπάρχει και σύγχυση με το κόστος και τα λοιπά. Άρα λοιπόν πιστεύουμε πως είναι σκόπιμο να υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες αλλά με βάση την πραγματική απόδοση, ώστε να αποφεύγεται αυτό το ζήτημα, το, πρόβλημα της ανυπαρξίας αυτών των δεδομένων. Αλλά θέλω να τονίσω και πάλι ότι δεν είναι το βασικό ζήτημα που μας απασχολεί όσον αφορά την απόδοση. Το βασικό ζήτημα που μας απασχολεί είναι τα σενάρια που έχουμε αναφέρει, όπου μόνο εξετάζονται οι δυνατότητες να το έχουμε όλα αυτά σε συνδυασμό, ώστε να αποφύγουμε ότι αυτή η έλλειψη πληροφορίας υπά, να, να, να, συνεχίσει να επικρατεί. Now, in terms of um, the multi-investment Όσον αφορά τις ε, επιλογές, πολυ, τις πολυεπενδυτικές επιλογές. Θα πρέπει να έχουμε μια λύση στο σχέδιο RTS. Η εταιρεία κάθε φορά θα πρέπει να διαθέτει τις πληροφορίες με βάση αυτό το πακέτο PRIP. Εάν υπάρχει ας πούμε μια ασφαλιστική εταιρεία που πολλά με διάφορα, ένα συνδυασμό διαφόρων ε, ασφαλιστικών ταμείων, επενδυτικών ταμείων, θα πρέπει να μπορεί να εξασφαλίσει τις πληροφορίες στον μελλοντικό της πελάτη για τα διάφορα επενδυτικά ταμεία στα οποία επενδύουν. Βέβαια υπάρχει και το θέμα της σχέσης με τα όσα αναφέρει η και την υποχρέωση των επενδυτικών ε, ταμείων να χρησιμοποιούν αυτήν την νομοθεσία. Πάντως πιστεύουμε πως τελικά αυτό που έχει σημασία είναι οι πληροφορίες που παίρνει ο καταναλωτής όταν ας πούμε η ασφαλιστική εταιρεία του παρέχει αυτήν την συμβουλή για επένδυση σε κάποιο συγκεκριμένο ταμείο. Θα πρέπει να υπάρχουν πρακτικοί τρόποι να εφαρμόζονται όλα αυτά με τρόπο ώστε καθώς περνά ο χρόνος να φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου τα παλιότερα, οι παλιότερες δέσμες θα μετατρα, μετατραπούν σε πρίψ. Υπήρχαν και κάποιες ερωτήσεις για τα παράγωγα. Εξ αρχής ε, στην διαβούλευση έχουμε αποσαφενήσει ότι εδώ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα και αυτό προέκυψε και από τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Ήταν σαφές. Αυτό τώρα επί το οποίο εργαζόμαστε μετά τις διάφορες ε, διαβουλεύσεις είναι ότι προσπαθήσαμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες ε, για το πώς τα διαφορετικά είδη παραγόγων θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στα κριτήρια για την αποκάλυψη των στοιχείων. Και είμαι βέβαιος ότι στο τελικό έγγραφο το τελευταίο αρτίας που θα στείλουμε στην Επιτροπή θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες μετά από τις διαβουλεύσεις που γίνονται. Αλλά θα πρέπει να είναι σαφές ότι θα περιλαμβάνονται, βεβαίως. Τώρα, για τον δείκτη κινδύνου και το στοιχείο που αναφέρατε ότι θα πρέπει να είναι ένας ο δείκτης. Να τονίσω κάτι που πιστεύω όλοι πρέπει να λάβουμε υπόψη. Όλα αυτά τα κάνουμε για τους καταναλωτές. Και γι' αυτό και το Κοινοβούλιο τόσο πολύ ήθελε να δοκιμαστούν με τους καταναλωτές εντός αυτού του προγράμματος και το κάναμε αυτό. Και μάλιστα ένα από τα πορίσματα, τα πιο σημαντικά πορίσματα ακριβώς αφορά αυτό το πεδίο Μα τη λέει ότι για να καταλαβαίνουν οι καταναλωτές καλύτερα θέλουμε έναν μόνο δείκτη και όχι διάφορους δείκτες που μετά μπερδεύουν τον κόσμο και δεν μπορούν να το αναλύσουν. Είναι εύκολο μήπως να περιλάβουμε ας πούμε κάποιους, ε, να βάλουμε ας πούμε στον ίδιο δείκτη τον κίνδυνο της αγοράς και το κίνδυνο της πίστοση. Όχι, δεν είναι εύκολο. Έχουμε δοκιμάσει διάφορες μεθοδολογίε. Ε, η μεθοδολογία επί της οποίας εργαζόμαστε και τώρα την τελειοποιούμε πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει σε διαφάνεια. Θα λαμβάνει υπόψη βέβαια τα στοιχεία της επιθετικότητας αλλά και το, την μέγιστη πιθανή απώλεια, που, ζημιά που μπορεί να έχει κανείς επενδύοντας στο συγκεκριμένο μέσο και έπειτα υπάρχει εδώ ένα κάποιο παρεδόσε. Αλλά το πιο σημαντικό στοιχείο είναι να δώσουμε κάτι στον καταναλωτή που να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Και αυτό ήταν σαφές νομίζω στις δοκιμές για τους καταναλωτέ και πρέπει να ληφθεί υπόψη. Θα προχωρήσουμε με αυτό το δίκτυο στις κατηγορίες 1 μέχρι 7. Θα πάμε βέβαια βαθύτερα όσον αφορά τη μεθοδολογία, ώστε να είμαστε πιο σαφείς και πιο διαφανείς για το πόσο ομαδοποιούνται οι διάφοροι, τα διάφορα είδη κινδύνου, αλλά πιστεύω πως προς χάρη διαφάνειας και, και κατανόησης του καταναλωτή, αυτός είναι ο τρόπος να προχωρήσουμε. Για το κόστος και τη μείωση της απόδοσης, ε, να πω ότι θέλουμε να περιλάβουμε το νομισματικό και το ποσοστό ποσοστιαίο στοιχείο, αυτό ήταν μια ερώτηση και επίσης ε, για να είμαι πολύ σαφής θα έχουμε και έναν δείκτη συνολικού κόστους και αυτό το ρωτήσατε accumulation. Ah, yes, Α, ναι, το σωρευτικό κόστος θα έχουμε. τη συσσόρευση, την ομαδοποίηση όλου του κόστου. Νομίζω πως απάντησα σε ερωτήσεις. Αν όχι, ευχαρίστως. Ναι. Γκαμπριέλ, μια ερώτηση για να καταλάβω αυτό που ανέφερες για τα παράγωγα και είπες ότι θα έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Ανεφέρθηκε στη δυνατότητα ενός κατάλληλου kit πακέτου για αυτά μόνο. Μήπως μπορείς να μας πεις δύο λόγια παραπάνω. Η βασική ιδέα και αυτό είναι κάτι το οποίο αυτή την εβδομάδα μας απασχολεί είναι να συμπεριλάβουμε ε, τα βασικά στοιχεία του ΚΙΤ για τα ΠΡΙΠ και να δούμε πώς σε διαφορετικές μορφές παραγόγων μπορεί κανείς να εκπληρώσει τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στα ΚΙΤ. Βέβαια θα πρέπει να υπάρξουν πάρα πολλές λεπτομερείς εξηγήσεις για το ποια θα είναι αυτά τα είδη των παραγόγων τα οποία μπορεί να λειτουργήσουν με τον τρόπο αυτό. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για το χρονοδιάγραμμα νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να εμείνουμε στα αυτά που έχουμε συμφωνήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί ε, να μειώσει και το χρόνο μετάφρασης ε, και άλλες διοικητικές καθυστερήσεις να τις συρρυκνώσει. Έτσι ώστε πριν από το καλοκαίρι να έχουμε καταλήξει κάπου και να έχετε χρόνο κι εσείς για τις δυνατότητες παρέμβασης της ΕΙΟΠΑ. Θέλουμε το ταχύτερα δυνατόν να προχωρήσουμε για το ΙΜΠΑ και ΕΣΜΑ αυτό εξαρτάται από την εφαρμογή το MIFID επίπεδα 1 και 2 και δεν ξέρω τι θα γίνει για την εντολή για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά standards. Είμαστε στην φάση προετοιμασίας του κειμένου αυτού, θα αποσταλεί σε όλες τις επιμέρους αρχές και οι ίσα θα ε, διαβουλευθούν θα δουν τι επίπεδα γίνονται σεβαστά στην παρούσα φάση και μπορούν να επανέλθουν τώρα. Ε, τίθεται εδώ και το θέμα των στάνταρ σαν παράδειγμα του ΩΣΑ. Για το ΜΙΦΙΡ και ΜΙΦΙΔ, ένα-δύο. Εμείς πιστεύουμε ότι τα, κρύπ, τα πρίψα από τη μία και μιφιντ από την άλλη θα πρέπει να προχωρήσουν το καθένα ξεχωριστά. Δεν θα πρέπει να περιμένουν τα πρίψα επειδή καθυστερεί το μιφιντ και νομίζω ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να προετοιμάσουμε μια σωστή απάντηση στις ανάγκες ε, του ΚΙΤ. Και σύντομα σχόλια για το περιεχόμενο του ΚΙΤ. Αυτό φυσικά είναι υπό εξέταση από τη ΣΥΖΑ στην παρούσα φάση. Ε, οι προηγούμενες αποδόσεις σαν παράδειγμα. Νομίζω ότι βασικό είναι να δώσουμε χρήσιμα σενάρια στους καταναλωτές που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν τις δυνατότητες εξέλιξης των προγραμμάτων τους. Η συμπερίληψη των παλαιών αποδόσεων δεν είναι κάτι το απαραίτητο, αλλά δεν μπορεί να αγνοηθεί όταν να προετοιμάζουμε κάποια σενάρια, τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές επενδυτές για τα παράγωγα. Γνώμη μας είναι ότι εντάσσονται στο πρίψ. Δεν χρειάζεται να εξαιρεθούν. Το θέμα είναι να βρούμε έναν τρόπο πρακτικά να τα συμπεριλάβουμε και να μην χρειάζεται να υπάρχει συστηματική ενημέρωση η οποία να μην αποτελεί ρεαλιστικό βάρος για τους προτείνοντες μια τέτοια Τώρα τα προϊόντα πολλαπλών επιλογών, τα multi-options. Ε, είμαστε σε μεταβατική ε, φάση για τα usage και θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ό,τι εντάσσεται στα πλαίσια του PRIPS να είναι συγκρίσιμο. Ο προηγούμενος ομιλητής εξήγησε ότι αυτός ο οποίος παράγει ένα συνδυασμένο προϊόν θα πρέπει να ενημερώνει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να δημιουργείται ένα kit το οποίο να καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της επένδυσης. Σας ευχαριστώ. Έχουμε λίγο χρόνο. Αν ε, η συγκήτρια ή εν πάση περιπτώσει η αναπληρώτρια της συγκήτριας ή οι θέλουν να πάρουν το λόγο, να ζητήσουν κάποια διευκρίνηση, Ευχαριστώ. Όχι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ που ήλθατε. Σας ευχαριστώ για την ε, παρουσίαση. Σας ευχαριστούμε και για αυτά που είπατε για το χρωμοδιάγραμμα και για τη δουλειά που κάνετε. Για να αξιολογηθούν καλύτερα οι ιδιαιτερότητες κάποιων συγκεκριμένων προϊόντων μεταξύ των οποίων και τα παραγωγά. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Σα ευχαριστώ. Να διακόψουμε μέχρι τι 11 και 4. όπου θα γίνει η επίσημη ακρόαση με την υποψηφία για την θέση του εκλεκτικού διευθυντή της ΑΙΟΠΑ. Ευχαριστώ και διακόπτω τη συνεδρίαση.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 Dear colleagues, I think that we can start. Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Στο 7 τη ημερήσια διάταξη για την ε, διορισμό του νέου εκτελεστικού διευθυντή τη ΕΙΟΠΑ. Έχουμε λοιπόν ε, μια δημοσία ακρόαση σήμερα στο πλαίσιο του διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή της ΕΙΟΠΑ. Ανοιχτή διαδικασία επιλογής, ο κύριος Φάουστο Παρέντε, τον οποίο και ορίζω που έχει επιλεχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, από το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΙΟΠΑ για τη θέση αυτή και όπως γνωρίζετε και όπως ξέρετε υπόκειται σε ε, συνένεση του Κοινοβουλίου. Έχουμε λοιπόν την ακρόαση με τον ε, επιλεκτέντα υποψήφιο για τα επόμενα χρόνια. Για να επιβεβαιώσουμε τον κύριο Παρέντε και το Μάρτιο του 2016 θα ψηφίσουμε στο Στρασβούργο. Καλώς ήρθατε κύριε Παρέντε και θα σας δώσω πάρα αυτά το λόγο για να κάνετε τα εισαγωγικά σας σχόλια. Πέντε λεπτά και μετά θα έχουμε το γύρο ερωταπαντήσεων. Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ αξιότιμα μέλη τη Ευρω... ΕΚΟΝ. Θα ήθελα να σα πω καταρχάς ότι είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα στο σώμα που εκπροσωπεί άμεσα του Ευρωπαίου πολίτε. Να πω δύο λόγια για τι βασικέ προκλήσει που πιστεύω ότι θα έχουμε στον από τα επόμενα πέντε χρόνια και να πω και δύο λόγια για πώ σκοπεύω να συμβάλλω η αποστολή της ΕΙΟΠΑ είναι να συνεχίσει να ε, οικοδομεί αξιόπιστες εποπτικές αρχές. Τρεις προτεραιότητες έχουμε τα επόμενα πέντε χρόνια για τη σύγκληση, ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή και χρηματοπιστική σταθερότητα. Ενίσχυση αυτής. Φυσικά, τώρα έχουμε το Solvency 2 που έχει τεθεί σε εφαρμογή. Είναι πολύ καλή λοιπόν η ευκαιρία να αυξηθεί η σύγκληση μεταξύ των εθνικών προσεγγίσεων. Έχουμε περάσει από τη ρύθμιση στην εποπτεία και στη συγκλήση πλέον για να υπάρχουν οι όροι ανταγωνισμού και ίδια προστασία για όλη την Ευρώπη. Και πολλά έχουν γίνει προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά θα πρέπει πολλά ακόμα να γίνουν για να φτάσουμε στο επίπεδο της πλήρους εναρμόνιση. Έχουμε λοιπόν τα εργαλεία στη διάθεσή μα για να το πετύχουμε αυτό. Θα ήθελα να τονίσω ότι έχουμε ένα εγχειρίδιο για την εποπτεία, της σχετικές αναθεωρήσεις και τον ειδικό ρόλο τη ΕΙΟΠΑ για feedback αξιόπιστο και ανεξάρτητο προ τι εθνικές αρχές σε ό,τι αφορά τι τρέχουσες τους. Είναι σε μοναδική θέση η ΕΟΠΑ Έχει επισκόπηση των πρακτικών αυτών, μπορεί να τις θέσει ένα αμφιβόλο και να παρέχει συστάσεις για το τι είναι το πλέον κατάλληλο σε όλη την Ευρώπη. Δεύτερη προτεραιότητα, προστασία του καταναλωτή. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Αυτό αποτελεί βασικό στόχο. Προαπαιτείται λοιπόν να βελτιωθούν οι κανόνες για την ε, συμπεριφορά στην αγορά. Και εποπτεία, παρακολούθηση. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια αποτελεσματική ε, διαχείριση των προϊόντων, διανομής ε, με τις σωστές ρυθμίσεις, προκειμένου να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του καταναλωτή ενημερωμένες ε, πολιτικές. Για να πετύχουμε το στόχο λοιπόν αυτό, η σχετική οδηγία για την ε, εφαρμογή είναι κρίσιμη σημασία και η προ την κατεύθυνση λοιπόν αυτή κινείται βάσει και τη αρχή τη αναλογικότητα για την βελτίωση τη εναρμόνιση σε όλη την Ευρώπη. Με παράλληλο σεβασμό εκ παραλλήλου των διαφόρων των εθνικών αγορών και των διαφορών δικτύων κατανομής, διανομής. Συγγνώμη. Η βασική αρχή θα πρέπει είναι να καταλάβουμε κατά πόσον είναι ικανοποιημένο ο καταναλωτή και ποιε είναι οι ανάγκε του. Χρειάζεται λοιπόν προστιθέμενη αξία των προϊόντων για τον καταναλωτή και θα πρέπει να ξανακερδίσουμε λοιπόν, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του καταναλωτή για το τρίτο ζήτημα, για τους όρους της αγοράς. Ξέρουμε ότι τα ασφαλιστικά και συνταξιδετικά ταμεία ελέγχονται διαρκώ. Έχουμε αναπτύξει πολλά stress test, ε, δοκιμέ τέτοια αντοχή για να αντιμετωπίσουμε τα ασθενή σημεία. Θα συνεχίσουμε προ την κατεύθυνση αυτή λοιπόν για να υπάρξει και μια κοινή βάση δεδομένων στον τομέα των ε, ασφαλιών που θα επιτρέψει να βελτιωθούν οι δράσει μα και να συντονιστούν οι δράσει follow-up από πλευρά των εθνικών αρχών. Έχουμε και άλλα σημαντικά έργα. Αναθεώρηση του Solvency 2, του BED πανευρωπαϊκό συνταξιδοτικό πρόγραμμα, Global Capital Standards για τις ασφάλειες, η εφαρμογή του IRP και πάρα πολλά τέτοια project. Για να τα πετύχουμε λοιπόν αυτά, θα πρέπει να αλλάξει ο ΕΙΟΠΑ για να προσαρμοστεί στις ε, νέες μελλοντικέ φάσεις και προτίθεμαι να διαχειριστώ αυτές τις προκλήσεις και να φροντίσω η στρατηγική να μεταφραστεί σε καθημερινές, η σε καθημερινές δράσεις. Έχω μακρά εμπειρία σε διαχείριση τέτοιων περίπλοκων project. Εδώ και χρόνια εργάζομαι σε διεθνή περιβάλλον. Έχω σαφή ευρωπαϊκή νοοτροπία και υποστηρίζω ένθερμα την ευρωπαϊκή ιδέα. Προσφάτως η διαπραγμάτευση του IMDB βελτίωσε τις δυνατότητες παρακολούθησης των σχετικών διαδικασιών και την εξέβρεση λύσεων προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα άλλο project, η κατάρτιση του ΙΒΑ στην Ιταλία, με, μου επέτρεψε να βελτιώσω τις σχετικές διευθυντικές μου ικανότητες. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι θα ήταν μεγάλη μου τιμή να υπηρετήσω τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εάν επιλεχθώ για τη θέση αυτή προκειμένου να δημιουργηθεί και μια ισχυρή και αξιόπιστη υποπτική αρχή στο επίκεντρο έχοντας πάντα το συμφέρον του Ευρωπαίου πολίτη. Και φυσικά θα είμαι στη διάθεσή σας να αναφέρω οτιδήποτε χρειαστείτε ανά πάσα στιγμή. Και φυσικά λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ευρωπαϊκές α, Αυτά. Ευχαριστούμε τον κύριο Πάνη. Ευχαριστώ. Μπάλτς, ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Παρέντε, πολύ χαιρόμαστε που βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Δύο ερωτήσεις έχω να σας απευθύνω. Και ενδεχομένω να έχω και την ευκαιρία να δευτερολογήσω να κάνω και ερωτήσεις. Κύριε Παρέντε, ήσασταν τμήμα της δομής ΣΕΟΠΣ και στην, από την αρχή εκπροσωπούσασταν στο, στον ΕΙΟΠΑ. Συμμετείχατε στον ΕΙΟΠΑ. Πώς θα είσαστε λοιπόν αντικειμενικός και ανεπηρέαστος σε αυτή την ε, νέα σας θέση ως εκτελεστικός διευθυντής της ΕΙΟΠΑ και πώς ε, θα φροντίσετε να λεφτούν υπόψη οι αξιώσεις του Κοινοβουλίου για την ε, καθορισμό προτεραιοτήτων στην λειτουργία του ΕΙΟΠΑ για παράδειγμα το θέμα της αναλογικότητας. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Για πάρα πολλά χρόνια εργαστήκατε για τις Ιταλικές Υποπτικές Αρχές. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τι περιμένετε από τους πρώτους ισολογισμούς Solvency 2 των Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Εταιριών και Πώς αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο του να ανοίξουν αυτοί οι κανόνες ε, για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να τηρηθούν στην τελική ανάλυση ή προθεσμίες ε, για την αναθεώρηση των ε, νομοθεσιών αυτών από τους νομοθέτες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπάλτ για το πρώτο σημείο που δείξατε. Θα ήθελα να πω ότι ε, επί σειρά ετών εργάζομαι στο διεθνές, ε, στη διεθνή αγορά σε διάφορες θέσεις και συμμετείχα σε διάφορες θέσεις και στον ΕΙΟΠΑ και προφανώς έχω ξεκάθαρη ευρωπαϊκή νοοτροπία. Πάντα προσπάθουσα να βρω μία λύση και να ξεπεράσω τα εμπόδια υπέρ του ευρωπαϊκού project, υπέρ των ευρωπαϊκών εξουσίων και αυτό νομίζω ότι το αναγνωρίζουν όλοι μου οι συνάδελφοι. Δεν πιστεύω ειλικρινά ότι τίθεται θέμα ανεξαρτησίας και ασφαλώς κατευθυντήρια γραμμή μου θα είναι να μεταφραστεί η στρατηγική του ΕΙΟΠΑ σε μια καθημερινή δραστηριότητα, σε μια καθημερινή δραστηριότητα με την έγκριση και των κοινοβουλίων και των ε, υπόλοιπων θεσμικών οργάνων. Δεν πιστεύω ότι τίθεται θέμα κριτική στο σημείο αυτό. Για το δεύτερο ζήτημα, φυσικά και πρέπει να θεωρήσουμε. Κανένα project, ε, ξέρετε, δεν είναι τέλειο. Το Solvency 2 αναπτύχθηκε μετά από κάποια χρόνια. Και ήδη τώρα δημιουργείται σε κάποιε περιπτώσει εντύπωση ότι είναι υπερβολικά πολύ σύνθετο. Συμφωνώ. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην αναθεώρηση του Solvency 2. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι θα πρέπει να ισχύουν οι γενικοί κανόνε και μετά να δούμε ποιοι είναι οι τομεί όπου θα πρέπει να αναθεωρηθεί το σύστημα. Αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Yeah, you make a follow-up. You... Μια δεύτερη ερώτηση. Πείτε μας δύο λόγια για την αναλογικότητα. Για την αναλογικότητα έχουν γίνει ήδη αρκετά πράγματα μέχρι τώρα, ιδιαίτερα στον τομέα της ε, δημοσιοποίησης των στοιχείων. Θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια. Αναλογικότητα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν πράγματα αλλά είναι δική μας αρμοδιότητα να εντοπίσουμε σωστά τους τομείς στους οποίους η αναλογικότητα πρέπει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Ακόμα και σε επίπεδο θεμάτων προστασίας του καταναλωτή πρέπει να προσπαθήσουμε να μην υπάρξει μια αν θέλετε φυγή προς τις μεγαλύτερες γενικά μονάδες Πάντως ε, και στα πλαίσια της διακυβέρνησης κάποια πράγματα έχουν γίνει και εξακολουθεί να υπάρχει χώρος για ανάπτυξη της ε, αναλογικότητας. Δεν ξεκινήσαμε από μια τέλεια κατάσταση, θα πρέπει να βιώσουμε το περιβάλλον του Solvency 2 και να δούμε στα πλαίσια του Solvency 2 ποιες είναι οι δυνατότητες τις οποίες έχουν ενημερώνουμε σωστά τους εμπλεκομένους, έχουμε τα μέσα και νομίζω ότι μπορούμε να παίξουμε ηγετικό ρόλο. Φερέιρα έχει το λόγο. Κύριε Παρέντε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στην Επιτροπή μας. Θα μιλήσω κι εγώ αγγλικά διευκολύνοντας τον διάλογο, λέει η κυρία Φερέιρα. Ζούμε καιρούς ενδιαφέροντες αλλά και επικίνδυνους παράλληλα. Η ΑΙΟΠΑ είναι ένα νέο αν θέλετε όργανο, είναι μια νέα αρχή αλλά έχει πάρα πολλές ήδη σε εισαγωγικά ενοχλήσεις ε, για τον προϋπολογισμό της. Θα πρέπει και εσείς λοιπόν σύντομα να προχωρήσετε σε κάποιες επιλογές. Αυτή είναι και η ερώτησή μου η πρώτη. Αν πρέπει να επιλέξετε κάποιους τομείς της αρμοδιότητάς σας, ποια είναι η άποψή σας για το τι πρέπει να κάνει η ΑΙΟΠΑ. Θα συμπεριλάβετε το θέμα της προστασίας των καταναλωτών. Δεύτερον, θα πρέπει να ενισχύσουμε, καλούμεθα να ενισχύσουμε τους δεσμούς ανάμεσα στις διαφορετικές εποπτικές αρχές, γιατί στο εσωτερικό των χρηματαγορών δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στις διάφορες μορφές δραστηριότητας. Πώς θα διασφαλίσετε εσείς την συνεκτικότητα και την συμβατότητα του πλαισίου λειτουργίας της ΙΑΙΟΠΑ με άλλα όργανα, άλλες αρχές. Και τέλος, κάτι το βασικό για τους καταθέτες, τους αποταμιευτές μάλλον, είναι να κατανοήσουν σωστά τους κινδύνους στην ασφαλιστική αγορά και να δούνε ακριβώς πώς κάποια προϊόντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να συγκεντρώσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και να μπορέσει κανείς να, εμπιστευθεί τις καταθέσεις του σε τέτοιου είδους προϊόντα χαμηλής απόδοσης βέβαια. Έχετε δίκιο εμείς ε, βιώνουμε καιρούς ενδιαφέροντες και δύσκολους. Συνολικά σαν χρηματοπιστωτικές αγορές πρέπει να βάλουμε κάποιες προτεραιότητες. Ξεκινάμε από την προστασία των καταναλωτών. Όλες οι δράσεις μας συνδέονται με την προστασία των καταναλωτών. Οι προτεραιότητες λοιπόν είναι απαραίτητο να καθοριστούν, ιδιαίτερα όταν σε δημοσιονομικό επίπεδο δεν έχουμε επαρκή μέσα και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξή του ε, για τον προϋπολογισμό μας. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτό και στο μέλλον. από την άλλη <coughs> πρέπει να αντιμετωπίζουμε το θέμα ε, της ε, έλλειψης πόρων. Ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε streamlining των διαδικασιών μας, αλλά η προστασία των καταναλωτών είναι κομβική για μας και θα συνεχίσει να είναι. Νομίζω ότι έχουμε τις δυνατότητες να κάνουμε καλές προτάσεις, καλούς σωστούς κανόνες, και να ε, επιβλέψουμε σωστά τον τομέα αυτό και με θεματολογικές ε, ε, εκθέσεις μέσω των στοιχείων τα οποία μπορούμε να συλλέξουμε να επιλέξουμε έτσι μεθόδους αναφοράς που βελτιώνουν την προστασία του καταναλωτή. Για τη συνεργασία με τις άλλες εποπτικές αρχές Νομίζω ότι η κοινή ε, επιτροπή δουλεύει καλά. Εγώ ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής των Υπευθύνων για τις Επιμέρους Αρχές και υπάρχει ανάγκη για την βελτίωση της συνεργασίας αυτή σίγουρα, αλλά υπάρχει ένα σωστό πνεύμα συνεργασίας, απαιτείται αμοιβαίος σεβασμός, αναγνώριση των διαφορών ανάμεσα στις διάφορες αρχές και τομείς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να συνεργαστούμε. Για το ΠΑΠΣ νομίζω ότι αυτά τα ασφαλιστικά προγράμματα σε ταμεία συνταξιοδοτικά ευρωπαϊκού επίπεδου είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά ελκυστικό. Μέχρι τώρα έχουμε περισσότερο εθνικές αγορές και όχι σε επίπεδο εσωτερικής αγοράς συνολικά. Θα υπάρξει δυνατότητα βελτίωσης των δυνατοτήτων των καταναλωτών έτσι ώστε ε, να βοηθήσουμε και εμείς την χρηματοδότηση του συστήματος ε, του ασφαλιστικού. Ε, βρισκόμαστε στην φάση της διαβούλευσης, συλλέγουμε τα σχόλια των χρηστών και νομίζω ότι θα σας ενημερώσουμε σύντομα. Ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε. Ο συνάδελφος Καθηγητής σα ε, σας σε διάφορες ερωτήσεις σε προηγούμενες ε, ακροάσεις. Θέλω όμως ε, να ε, σας ρωτήσω κάτι για τα εποπτικές αρχές και το ρόλο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με το Κοινοβούλιο. Έχουν περάσει διάφορες νομοθεσίες από την ίδρυση των ε, εποπτικών αρχών, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν κάποιο είδους δευτερεύοντες κανόνες και ο ρόλος μεταξύ των εποπτικών αρχών και της Κομισιόν όταν σχημάτισαν το RTS. Αυτό μας απασχολεί και αυτή η η, η, η τριγωνική συζήτηση είναι προβληματική. Η, ο δημοκρατικός έλεγχος ε, του επίπεδου 2 είναι εξαιρετικά σοβαρός. Οπότε το ίδιο είναι και ο διάλογος, ο συνεχιζόμενος διάλογος ανάμεσα σε ευρωπαϊκές αρχές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διάρκεια της διαδικασίας επίπεδου 2. Εσείς προσωπικά πώς θα εξασφαλίσετε ότι η ΟΠΑ θα διαβουλεύεται πλήρως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν υιοθετήσει μέτρα δεύτερου επίπεδου, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες εμείς να το περιορίσουμε στο μέλλον. Και έπειτα με την εθνική σας εμπειρία θα εξασφαλίσετε την συνεπή εφαρμογή από τους εθνικούς επόπτες για μέτρα όπως τα μέτρα της Solvency 2. Σας ευχαριστώ. Κατάρχά. ναι, υπάρχει ανάγκη να φτιαχτεί η δευτερεύουσα νομοθεσία, γιατί όλες οι λεπτομέρειες δεν μπορούν να ρυθμιστούν στο πρώτο επίπεδο. Αυτό νομίζω είναι σαφές. Επίσης πρέπει να είμαστε ε, υπόλογοι, να λογοδοτούμε και να ερχόμαστε να αποβάλουμε τις εργασίες μας κάθε φορά Ε, καθώς και να ακούμε τα αιτήματά σας, τις ανησυχίες σας και τα λοιπά. Και βεβαίως ε, και δεσμεύομαι να βρίσκω χρόνο οποτεδήποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο ώστε να μπορούμε να συνομιλούμε και να διαβουλευόμαστε. Για μένα είναι σαφές ότι υπάρχει σαφής ανάγκη για λογοδοσία και για ε, παρουσίαση των εργασιών μας κάθε φορά. Ως προς αυτό ίσως ένα ακόμα βήμα θα μπορούσε να είναι μία συνεργασία μεγαλύτερη στη διάρκεια της ανάπτυξης του πρώτου επίπεδου με τις ε, εποπτικές αρχές της ΕΖΑ για να καταλάβουμε καλύτερα ε, ποιοι είναι οι τομείς όχι ποιο είναι ο τομέας των συνομοθετών, αλλά για να καταλάβουμε καλύτερα ποια είναι η λογική που διέπει κάποιες διατάξεις του πρωτογενούς, ε, της πρωτογενούς νομοθεσίας και έτσι να μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω ε, τις εργασίες υπό την έννοια της νομοθεσίας ε, του επίπεδου 1. Για μένα ο διάλογος είναι απαραίτητος σε όλες τις φάσεις των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Μέχρι στιγμής ε, δεν γινόταν στο δεύτερο επίπεδο. Νομίζω έχουμε ε, μια ανεξαρτησία από την Κομισιόν όταν συντάσσουμε τις ε, συμβουλευτικές μας γνωμοδοτήσεις. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις δικές σας επιθυμίες και αιτήματα. Ένα τομέας περαιτέρω βελτίωσης κατά από αυτό που κατάλαβα είναι το να μπορείτε να ακούσετε από εμά πότε αναπτύσσετε το πρώτο επίπεδο για να καταλάβουμε καλύτερα ποιο είναι το λογικό πίσω από όλα αυτά. Ποια είναι η λογική. Και, ε, και έτσι θα είναι πιο ομαλή η λεπτομερής εφαρμογή στο επίπεδο 2, 3 κτλ. και στο εθνικό επίπεδο για το Solvency 2 και την εφαρμογή των νομοθεσιών. Και εμεί συμμεριζόμαστε τι ανησυχίε των υπολείπων χωρών γιατί η Solvency 2 από όσο έχω ακούσει είναι ριζική αλλαγή και βεβαίω φέρνει μαζί της ευκαιρίε αλλά και φόβου. Υπήρξε έτοιμα για να έχουμε λεπτομερείς οδηγίες για το πώς να εφαρμόσουμε το νέο σύστημα. Επ' αυτού ήταν πολύ βοηθητικό το ότι αναπτύξαμε σε επίπεδο ΙΟΠΑ τις ε, κατευθύνσεις γραμμές που αναπτύξαμε. Αν και κάποιες φορές είναι υπερβολικά πολλές, αλλά πάντως βοήθησαν στο να δώσουν λεπτομερείς απαντήσεις και με εναρμονισμένο τρόπο στις ε, Ιταλικές ασφαλιστικές εταιρείες, γιατί διαφορετικά θα είχαμε ακόμα περισσότερα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιάτσεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κόρα μου έδωσε 87 ερωτήσεις, αλλά θα θέσω μόνο κάποιες από αυτές. Κύριε Παρέντε, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα πιο σημαντικά συμπεράσματα στα οποία καταλήξατε τα τελευταία τρία χρόνια στην παρούσα εργασία σας και τι εμπειρία έχετε να προσθέσετε στην ΙΑΙΟΠΑ. Και δεύτερον, τι αλλαγές θα κάνετε στην καθημερινή διαχείριση της ΙΑΙΟΠΑ, αν κάνετε. Και πώς οι αλλαγές αυτές θα βελτιώσουν τη λειτουργία της. Και τέλος, ποιες είναι οι πιο μεγάλες δυσκολίες και προκλήσεις για την ΙΑΙΟΠΑ τα επόμενα πέντε χρόνια, εσωτερικές και εξωτερικές. Thank you. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας, για την πρώτη σας ερώτηση. Εγώ έχω μία εμπειρία ιδιαίτερα στον τομέα των αλλαγών. Τα τελευταία τρία χρόνια σημειώνω την εξέλιξη της εθνικής μου αρχής. Υπήρξε μια μεταρρύθμιση τα τελευταία χρόνια που επέτρεψε στην ελεγκτική μου αρχή να αποκτήσει νέα χαρακτηριστικά. Ήμουν υπεύθυνο για την Task Force στην οποία συμμετείχαν ε, και παλαιοί εκπρόσωποι της Εποπτικής Αρχής και εκπρόσωποι της Κεντρικής Ιταλικής Τράπεζας. Στην Ιταλία, όπως ξέρετε, υπήρξε μια συγχώνευση της Εποπτικής Αρχής για τα πιστοτικά ιδρύματα με την αντίστοιχη Εποπτική Αρχή ε, για τα ασφαλιστικά ιδρύματα. Εμείς προσπαθήσαμε λοιπόν να ενιοποιήσουμε την διαδικασία μέσω της νέας κατανομής πόρων και δημιουργήσαμε και ένα νέο οργανόγραμμα. Όλες αυτές οι εμπειρίες νομίζω ότι είναι σημαντικές για την ΙΑΙΟΠΑ. Και εδώ έρχομαι στη δεύτερη ερώτησή σας γιατί και η ΑΙΟΠΑ βρίσκεται στην ίδια περίπου κατάσταση. Έχει αναπτυχθεί τον τελευταίο καιρό, έχουν πετύχει πολλά τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά νομίζω τώρα εφόσον περνάμε από την ρυθμιστική λειτουργία στην εποπτική λειτουργία, απαιτείται ίσως μια αλλαγή της ε, προσπάθειας που γίνεται. Πρέπει να υπάρξει μια σωστότερη εκπαίδευση του προσωπικού για την εφαρμογή της πολιτικής μας και θα πρέπει ε, εμείς να ασχοληθούμε κυρίως με το θέμα της εποπτικής σύγκλησης, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρξει νέα κατανομή τμήματος του προσωπικού. Λοιπόν, η Ιταλική μου εμπειρία σύνεπως μπορεί να είναι καποφόρα και στη συγκεκριμένη αυτή προσπάθεια για τα επόμενα πέντε χρόνια. Τώρα για τις δυσκολίες της ΑΙΟΠΑ, για τις εξωτερικές δυσκολίες, νομίζω ισχύουν για το σύνολο των ασφαλιστικών ε, γενικά ε, τομέων. Η χρηματοοικονομική κατάσταση, οι θέσεις των ασφαλιών, των ασφαλιστικών μάλλον ταμείων αντιμετωπίζουν πολλά θέματα. <clears throat> Συνεχίζουμε να προχωράμε στα stress test, στα τεστ αντοχής για να εντοπίσουμε τα εύθραυστα στοιχεία και να επιτρέψουμε στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να αναλάβουν δράση και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε στο μέλλον κάποιες εξωτερικές συνθήκες, συνθήκες αγοράς να δημιουργήσουν κρίσεις. Έχουμε τα απαραίτητα μέσα, πρέπει με τα μέσα αυτά να δουλέψουμε. Το Solvency 2 θα μας δώσει και μία βάση δεδομένων για τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και θα μπορέσουμε έτσι να βελτιώσουμε τις ικανότητές μας για τον εντοπισμό των ευάλωτων σημείων μας και να υπάρξει δυνατότητα παρέμβασης προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ε, δεν υπάρχει εκπρόσωπος της ΓΟΥΕ, Περνάμε στους πρασίνους. Ο Σβέν Γκίγκολντ έχει το λόγο. Καλώς ορίσατε και καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι σας ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε εδώ σήμερα και είναι σαφές ότι οι, οι ικανότητες σας προκύπτουν από το βιογραφικό σας, είστε καλά προετοιμασμένος ε, για τη δουλειά αυτή. Ωστόσο, ο ρόλος μας ως πράσινη είναι πάντα να κοιτάμε τα σημεία τα ευαίσθητα και να ασκούμε κριτική. Μην το πάρετε λοιπόν προσωπικά. Είναι ο ρόλος τον οποίο έχουμε προδιαγράψει εμείς για τον εαυτό μας εδώ. Στις διαπραγματεύσεις, το τελευταίο στάδιο του Solvency 2, είδαμε πολύ μεγάλη δραστηριότητα από πλευρά τη Ιταλική ε, κυβέρνηση για να υπάρξει ειδική αντιμετώπιση προ αυτήν. Δύο θέματα λοιπόν θα ήθελα να υπογραμμίσω. Σε ό,τι αφορά το πριν αντικυκλικότητα, ασύμετρο και το οποίο είναι κατά τη λογική του χρηματοοικονομικού κανονισμού κατά κάποιο τρόπο σε ό,τι αφορά δηλαδή την κίνηση των ε, αγορών προς τη μία κατεύθυνση και όχι προς την άλλη. Ασκήθηκε λοιπόν έντονη πίεση προς από την Ιταλική κυβέρνηση για το αντικυκλικό αυτό premium. Και κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά το lobbying της Ιταλίας για την ε, συμμετοχή στο Solvency 2, για την συμμετοχή των ασφαλιστών εξορισμού να είναι άνευ κινδύνου. Πείτε μας λοιπόν, συμμετείχατε. Συμμετείχατε στην διαδικασία λήψη αποφάσεων στην Ιταλία ε, για να υποστηριχθούν από πλευρά τη Ιταλική κυβέρνηση οι θέσει αυτέ, τι διαπραγματεύσει και κατά δεύτερον, ποια είναι η προσωπική σα άποψη για τα δύο αυτά θέματα, γιατί και τα δύο αυτά είναι κατά τη αρχή ε, του Solvency 2. την αρχή της πρόληψης. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Να σας πω ότι συμμετείχα ως τεχνικός, να σας το πω, ως εμπειρογνώμονας ε, στις διαπραγματεύσεις για το Solvency 2. Σύμβουλος του αρμόδιου Υπουργού. Και σε κάποιε περιπτώσεις ήμουν εκεί και στις συνεδριάσεις ε, στο Συμβούλιο για να εκπροσωπήσω την Ιταλική κυβέρνηση. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν τα σημεία αυτά τα οποία δείξατε τουλάχιστον σε κάποιες φάσεις ε, του project. Για το πρώτο θέμα που δείξατε, όντως μπορούμε να πούμε ότι το πριμ αντικυκλικότητα στο οποίο τελική ανάλυση δεν είναι αυτό που έχει εφαρμόσει πλέον η οδηγία Solvency 2 τότε η Ιταλία άλλα πράγματα έχει ζητήσει εν περιπτώσει σε τελική ανάλυση το τρέχον σύστημα σίγουρα δεν αντίκειται με την αρχή της ε, πρόληψης. Πρόκειται για ένα μέσο μόνο αντιστάθμισης σε κάποιες περιπτώσεις κρίσης και εμείς ασφαλώς θα πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς λειτουργεί όταν το εφαρμόζουμε. Ναι, ναι, ναι, ο κύριος Γκίκολ, επιτρέψτε μου να ρωτήσω. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, σας παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος, αφήστε τον να ολοκληρώσει και μετά ξαναρωτάτε. Όχι, όχι, δεν, δεν διακόπτουμε εδώ. Να ολοκληρώσει πρώτα. Ο υποψήφιος. Όπως σας είπα, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε ενδεχόμενε αλλαγές του συστήματος τραποποίησης σε περίπτωση που υπάρχουν ε, σημεία αδύναμα. Έχουμε εφαρμόσει λοιπόν ε, την πρώτο γύρο. Θα συγκεντρώσουμε ε, τις εμπειρίες από τα πρώτα έτη της λειτουργίας του και θα δούμε πώς θα τα βελτιώσουμε. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε συγκεκριμένα ποιες είναι οι δυναμίες του συστήματος για το δεύτερο θέμα, γιατί η συμμετοχή. Έχετε δίκιο. Δεν είναι άνευ κινδύνου η συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιριών. Υπάρχει ένας παράγοντας υπολογισμού χαμηλότερος, ένας συντελεστής μάλλον, χαμηλότερος από αυτό που χρησιμοποιούσαμε τότε, κατά το παρελθόν. Τότε, θεωρήσαμε ότι για μια τέτοια μακροπρόθεσμη επένδυση όπως είναι η συμμετοχή δεν είναι αντίθετη δεν είναι αντίθετο αυτό ο συντελεστή ε, με την αρχή τη πρόληψη του Solvand-Se 2. Φυσικά, μπορεί κανεί την αδιαφωνία, αλλά αυτή η απέτηση για μακροπρόθεσμη επέντιση σήμερα καθίσαμε κάτι σημαντικό. Και πιστεύω πραγματικά ότι ακόμα και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δείξουμε προσοχή σε ό,τι αφορά την αναθεότηση του Solvency 2. Φυσικά μπορεί κανει να διαφωνεί, αλλά αυτή η απέτηση για μακροπρόθεσμη επένδυση σήμερα καθίσταται κάτι σημαντικό. Και πιστεύω πραγματικά ότι ακόμα και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δείξουμε προσοχή σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του Solvency 2 για να δούμε κατά πόσο θα χρειαστεί να αλλάξουμε το συντελεστή υπολογισμού της συμμετοχής υποθέτω ότι θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Αλλά δεν πρόκειται να τις αποφασίσω εγώ εδώ και τώρα. Μάλιστα, follow-up. Ε, δευτερολογία. Ακόμα και αν δεν έχετε χρόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Το θέμα όμως είναι πολύ απλά ότι δεν καταλαβαίνω γιατί το πριμ αντικυκλικότητας δεν αντίκειται με την αρχή της ε, πρόληψης. Αποδέχεστε ουσιαστικά ότι οι τιμές μπορούν να πέσουν στις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά δεν αποδέχεστε τον σχηματισμό αποθεματικών. Κατά δεύτερον, δεν σας ζήτησα να πάρετε απόφαση, αλλά ζητάτε είστε υποψήφιος για μια θέση εδώ πρέπει να τοποθετηθείτε. Πείτε μας λοιπόν ποια είναι η άποψή σας για την ιδιωτική αυτή συμμετοχή. Και όταν είναι λογικό οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις να έχουν ιδιαίτερα πλεονόμια όταν είναι με τη μορφή συμμετοχή και όχι οι υπόλοιπε μακροπρόθεσμε επενδύσεις. Ναι, σα δίνουμε πολύ παραπάνω χρόνο, λέει ο Πρόεδρος από τα άλλα μέλη. Και δεν ξέρω, θέλετε να εφαρμοστεί ο κανονισμό ή θέλετε, εν πάση περιπτώσει, η απάντηση. Όπω είπα, καταλαβαίνω τι λέτε. Θα πρέπει να κατανοήσουμε πώ λειτουργεί το νέο σύστημα, γιατί το πρίμα αντικυκλικότητας δεν είναι ένα μόνο ενιαίο μέτρο. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων μακροπρόθεσμων, τα οποία αντισταθμίζονται ουσιαστικά από κάποιες ποιοτικέ απαιτήσει. Δεν είναι δεδομένο και σίγουρο ότι αποτελεί απλά μία μορφή παράλογης προσέγγισης του ζητήματος. Πολύ λυπάμαι, αλλά αυτό δεν ελευθεύει, δεν στέκει. Θα πρέπει το σύστημα να το θεωρήσουμε στο σύνολό του. Η εφαρμογή των μακροπρόθεσμων μέτρων θα πρέπει να εξεταστεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Και ο επόπτης έχει στη διάθεσή του όλα τα εργαλεία για να κατανοήσει και να αξιολογήσει κατά πόσο τα μέτρα αυτά απλά επιτρέπουν να ξεπεραστεί μια κρίσιμη στιγμή στην αγορά ή αποτελεί μια μη λογική, μη αναλογική προσέγγιση. Αυτή είναι άλλωστε η δουλειά, αυτό είναι το καθήκον του επόπτη. Μη φοβάστε λοιπόν. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Η FDD δεν υπάρχει κάποιος. Ούτε από το ENF. Οπότε επιστρέφουμε στον κύριο Μπάλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άλλη μια ερώτηση έχω να κάνω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρσι τον Νοέμβριο ανακοίνωσε ότι ε, πρόκειται να καταθέσει προτάσεις για περαιτέρω μείωση του ρίσκου, του κινδύνου και ότι αυτό θα ήταν προϋπόθεση για την ε, ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και των σχετικών διαπραγματεύσεων. Την περασμένη εβδομάδα ο Ματέο Ρέντσι ε, ανακοίνωσε ότι πρόκειται να προβάλλει βέτο κατά, κατά τον, του συστήματος αυτού για τα κρατικά ομόλογα. Και φαίνεται ότι όλα τα θεσμικά όργανα, η ΕΚΤ και το καθεξής, το εξετάζουν το θέμα αυτό. Πώς αξιολογείτε λοιπόν εσείς ε, την ε, δήλωση και διακήρυξη του κυρίου Ρέντσι και ποια είναι η προσωπική σας άποψη σε ό,τι αφορά τα κρατικά ομόλογα φαντάζομαι σε ό,τι αφορά τις ασφάλειες, όχι τις τράπεζες. Αστείο λέει ο πρόεδρος, αστείο. Κατανοώ αυτό που είπατε για τους κινδύνους σε επίπεδο χρέους. Νομίζω ότι στην παρούσα φάση δεν είμαστε σε θέση να έχουμε μία αντίληψη που λέγει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα έκθεσης κινδύνου σε σχέση ε, με το ευρύτερο χρέος. Υπάρχουν μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν και σε επίπεδο τραπεζικό και σε επίπεδο ε, ασφαλιστικό έτσι θα μπορέσουμε να δούμε τι λεπτομέρειες μπορούμε να έχουμε σε επίπεδο μακροπροληπτικό και μικροπροληπτικό. Αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο θα πρέπει να εργαστούμε και για την αναθεώρηση της Solvency 2 μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Για τον κύριο Ρέντσι, ο Πρωθυπουργό μου είναι ο κύριος Ρέντσι, μερικές φορές συμφωνώ με αυτά που λέγει, μερικές φορές λιγότερο. Αυτά. Νομίζω ότι ο διευθυντής της ΙΑΙΟΠΑ δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις οδηγίες του Πρωθυπουργού του, ευτυχώς. Κυρία Γκίλ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Παρέντε. Την προηγούμενη εβδομάδα η ΑΙΟΠΑ εξέθεσε τις προτεραιότητές της για το 2016. Just last year. Δεν υπήρξε θέματα για τα FinTax. Τα FinTax πάνε καλά. Υπήρξαν στο Ηνωμένο Βασίλειο επενδύσεις ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ. Μπορούν να αλλάξουν πολλά στον χρηματοπιστωτικό τομέα και όχι μόνο στις τράπεζες, αλλά και στις ασφάλειες. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κοινωνία που αλλάζει ε, συνεχώς σε τεχνολογικό επίπεδο η πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουν οι εποπτικές και αριθμιστικές αρχές είναι το πώς θα προσαρμοστούν καλύτερα σε αυτές τις αλλαγές και περιμένουν περισσότερα από τις υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να παρέχονται, θέλουν όλα να γίνονται καλύτερα, όλα θέλουν να γίνονται κυρίως όμως γρηγορότερα. Και πώς μπορούμε εμείς να διευκολύνουμε τη ζωή του καταναλωτού. Βλέπουμε λοιπόν κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες επιτρέπουν να, να αγοράζει κανείς μέσα σε δευτερόλεπτα αν είναι πολύ γρήγορος ασφαλιστική κάλυψη για το αυτοκίνητό του μόνο με μια φωτογραφική μηχανή και ένα τηλέφωνο φορητό, κινητό τηλέφωνο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε για να καλύψουμε λοιπόν αυτές τις τεχνολογικές αλλαγές που επαναλαμβάνω αλλάζουν τα τοπία που γύρω μας. Τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε ο τομέας αυτός να συνεχίσει να καλύπτει τις ανάγκες, να καινοτομεί αλλά χωρίς να υπαναχωρήσει ορισμένους τομείς. Πράγματι, είπατε ότι η τεχνολογία είναι αλήθεια, μας δίδει τεράστιες δυνατότητες, παρουσιάζει όμως και κάποιους νέους κινδύνους. Εμείς σαν εποπτική αρχή πρέπει να επιτρέψουμε στην αγορά να εκμεταλλευτεί τις νέες ευκαιρίες και να διασφαλίσουμε όμως ότι οι καταναλωτές, οι πολίτες αντιμετωπίζονται με προσοχή, χωρίς επιπλέον κινδύνους. Πώς θα γίνει αυτό είναι μερικές φορές εύκολο να επιβλέπει κανείς μια δεδομένη πλατφόρμα η οποία παρέχει ασφαλιστικά προγράμματα. Αν δει κανείς τον αριθμό των παραδοσιακών ενδιαμέσων που είναι σε επαφή με τον πολίτη, δεν μπορεί κανείς να είναι ανάμεσα στον ενδιάμεσο ασφαλιστή και τον πολίτη για να ελέγχει αν αυτά τα οποία λέγονται και η συμπεριφορά του ενδιαμέσου ε, είναι προς το συμφέρον του ασφαλιζομένου. Ε, γι' αυτό λοιπόν μια τεχνική πλατφόρμα είναι με βασική πηγή πληροφόρησης για τον επόπτη γιατί με μια χρήση της μορφής ελέγχου τότε μπορεί να συλλέγει τα στοιχεία που επηρεάζουν τα τεχνολογικά μέσα ε, που χρησιμοποιούνται όπως τα έξι τα τηλέφωνα. Έχουμε την δυνατότητα στην Ιταλία σαν παράδειγμα κάνουμε μία ανάλυση όλων των ιστοσελίδων σύγκρισης και πήραμε μέτρα εις βάρος αυτών που δεν ήταν συμβατά με τον κανονισμό. Έκαναν συγκρίσεις και αναλύσεις μόνο ανάμεσα σε ορισμένους ασφαλιστές οι οποίοι είχαν χρηματοδοτήσει άλλωστε την ίδια την ιστοσελίδα. Έχουμε λοιπόν τα μέσα να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις, αλλά σίγουρα τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα από ό,τι στο παρελθόν, στα πλαίσια της παραδοσιακής ασφαλιστικής αγοράς, όπου είχαμε απλά την παρουσία των ενδιαμέσων. Θα πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν να διασφαλίζουμε ότι οι κανόνες της αγοράς θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί ακόμα και αν παρέχονται μέσω ενός νέου τεχνολογικού μέσου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κλείσαμε τον γύρο των ομιλητών και τις ερωτοαπαντήσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει μία επιπλέον ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήμουν ε, μέλος της Επιτροπής ε, Εποπτείας των Ασφαλιστικών στην Ρουμανία και θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Παράντη καταρχάς και να ρωτήσω πώς προτίθεται να διαχειριστεί για παράδειγμα τις ε, ε, διαφωνίες μεταξύ των εθνικών αρχών όταν αυτές ανακύψουν τι είδους εργαλεία και μέσα θα χρησιμοποιήσετε και αυτό αποτελεί τροφή για σκέψη για όλους μας. Ξέρετε ότι στην παρούσα φάση ο ΙΟΠΑ κάνει μία μικροεποπτεία σε επίπεδο εθνικό, αλλά οι εθνικές ε, εθνικες οι αρχές διαφέρουν τόσο πολύ. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι οι εθνικές αρχές, ε, σε άλλες χώρες αυτό περιλαμβάνει τρία-τέσσερα διαφορετικά σώματα. Πιστεύετε ότι χρειάζεται να εφαρμόσουμε μια τυποποίηση ίσως του ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου σε εθνικό επίπεδο, γιατί αυτό θα απλοποιήσει τα πράγματα, θα υπάρξει καλύτερη σε εκπροσώπηση, συντονισμό και μεγαλύτερη απλούσταση, αν θέλετε, των πραγμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και έχετε δίκιο. Δεν μπορούμε απλά να τυποποιήσουμε τα πάντα. Δεν υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλους. Αλλά η σύγκληση, η σύγκληση σε θέματα εποπτεία είναι σημαντικό ζήτημα και θα πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Πρόκειται σαφώ για μία από τι προτεραιότητε τι οποίε έχουμε θέσει και όταν είπα ότι θα πρέπει να δούμε και να εξετάσουμε τις αρχέ αρχές εθνικό επίπεδο θα πρέπει να να συγκεντρώσουμε και να ενημερώσουμε όλη την Ευρώπη για τις βέλτιστες πρακτικές. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί μία και ενιαία και απλή προσέγγιση σε όλους. Όχι, θα πρέπει να λεφτούν υπόψη οι διαφορές στην αγορά, αλλά πιστέψτε με υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης της έξω κατάστασης σε ό,τι αφορά το επίπεδο εποπτείας. Σε ό,τι αφορά τη διαφωνία ενδεχομένω μεταξύ των εθνικών αρχών, προβλέπετε αυτό από την νομοθεσία και έχουμε τη διαμεσολάβηση ως αρμοδιότητα, μία από τις αρμοδιότητες του ΕΙΟΠΑ. Ελπίζουμε όλα αυτά να γίνουν χωρίς ε, να χρειαστεί καταφυγή στα τα μέτρα, αλλά αν χρειαστεί ο ΕΙΟΠΑ θα πρέπει να σε θέση να διαμεσολαβήσει μεταξύ δύο διαφορετικών εθνικών αρχών, μεταξύ και αυτό είναι ένα από τα μία από τις αρμοδιότητες που έχει χωρισία από τον νομοθέτη, από εσά προ τον ΙΟΠΑ και όπω σα είπα αυτό αποτελεί ένα μέσο ίσο της ανάγκη αν θέλετε, ίσο της προσφυγής για τις εθνικέ αρχές. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος, δεν βλέπω να ζητά κανείς άλλο το λόγο. Μπορούμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε την ακρόαση στο σημείο αυτό. σα ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παρέντα πολύ πολύ σύντομη α, συνεδρίαση κυκλισμένων των θυρών και στις 3.40 το απόγευμα θα γίνει σχετική ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ.